puhemies The sitting is open. Good morning, everyone. Καλημέρα σε όλους λέει η πρόεδρος. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Και αντίστοιχα